να υπάρχει τοπική <clears throat> απασχόληση και για μας και τις αναπτυσσόμενες χώρες και μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκρέζ για την Επιτροπή Απασχόλησης η κυρία Μπερέσ.